Συνάδελφοι, επειδή είμαστε πολυάριθμοι, σας παρακαλώ να κάνετε λίγη σιωπή για να ξεκινήσουμε. Για να επιτρέψουμε στην εισηγήτρια να λάβει το λόγο. Πρώτα απ' όλα έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Χθες σας στείλαμε μια νέα έκδοση της ημερήσιας διάταξης με ορισμένες τροποποιήσεις για τα θέματα που είχαν προβλεφθεί καταρχήν στις αλλαγές αυτές. Καταρχήν έχουμε την έκθεση για, την, για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που έχει παραπευθεί στην επόμενη Δευτέρα, επόμενη Δευτέρα, 27 Ιουνίου, δεύτερον, μετά από την απόφαση που ελήφθη στις 15 ε, Ιουνίου. Έχουμε και ένα σχέδιο ψηφίσματος για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΚΕΠΑ και ΕΠΑ. Τρίτο σημείο, προσετέθη η έκθεση του κυρίου Σάριους Βόλσκι για την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και τέλος έχουμε μια αντιπροσωπεία από το Μαρόκο και θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο συνταγματικής μεταρρύθμισης που, προ... που προτείνεται από τον ηγεμόνα του Μαρόκου. Και τέλος η ανταλλαγή με τον Αμίμπη Αλαράμπη, τον Υπουργό Εξωτερικών της ε, Αιγύπτου, ακυρώθηκε, γιατί όπως ξέρετε υπήρξε αναδιάρθρωση της κυβέρνησης στην Αίγυπτο. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν γίνεται δεκτή η ημερήσια διάταξη όπως έχει τροποποιηθεί. Ανακοινώσεις του Προέδρου βάσει της εντολής που εδόθη <clears throat> από το διευρυμένο Προεδρείο οι εισηγητές Μπροκ Γουαλτιέρη και Βερχόφστατ για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι δηλώσεις της υψηλής εκπροσώπου σε σχέση με την πολιτική ευθύνη της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και σε σχέση με τους τρόπους με τους οποίους θα λειτουργήσει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης στις εναρκτήριες φάσεις του με στόχο να συνταχθεί μια έκθεση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το φθινόπωρο του έτους αυτού και να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας και τις συστάσεις μας σε σχέση με τα θέματα αυτά. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στους ε, δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτρια είναι η κυρία Φρανσίσκα Καταρίνα Μπραντνερ. και θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο εκθέσεως. Η τροπολογία είναι η 17 Ιουνίου, λέει ο στις 12 η ώρα. Αυτή η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων λοιπόν έχει σημαντικό χαρακτήρα και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα λεγόμενα της κυρίας Μπράτνε. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που ήρθατε στις 9 για να ακούσετε τα περί δημοσιονομικού κανονισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης πρώτα απ' όλα για την συνεργασία μας, για τη γνωμοδότηση αυτή. Θεωρώ ότι βελτιώθηκε σημαντικά το κείμενο και θα ήθελα να τονίσω κάποια σημεία, όχι αυτά επί των οποίων όλοι συμφωνούμε. Τροπολογία 12, 11 και 4. Αυτά είναι τα τρία σημεία. Αρχίζω με την ε, τροπολογία 4. Ε, σας την παρουσίασα την περασμένη φορά, αν θυμάστε. Σε κάποιες ε, περιοχές ε, του κόσμου που δεν είναι στο φως δημοσιότητας καθημερινά, αναπτυσσόμενες χώρες, το Βαλού κτλ. Όπου έχουμε αντιπροσωπεία, αλλά δεν έχουμε πολύ προσωπικό από την υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης και αποφασίσαμε ότι μπορούν να ε, ε, μπορούν να εκχωρήσουν τον ναι, διαχείριση του προπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δούμε μέχρι το απόγευμα αν είναι δυνατόν να ζητήσουν άλλον επικεφαλής αντιπροσωπείας από άλλη χώρα που θα ε, έδινε την έγκριση γι' αυτό. Εάν είναι εφικτό, δεν χρειάζεται να αναπέμψουμε την αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό συνέστησε η κυρία Γκρέσλερ. Ε, είπε ότι αντί να επανεκχωρηθεί η αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή είναι μια καλή εναλλακτική λύση. Έτσι μπορούμε να έχουμε με καλύτερη χνηλασιμότητα για τα κονδύλια. Θα έχουμε αργότερα σήμερα την απάντηση. Ένα άλλο τώρα, ένα καταπίστευμα, καταπιστεύματα μάλλον, τροπολογία 11. Τα καταπιστεύματα Πιστεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η επικεφαλή ε, των ε, αντιπροσωπιών, αλλά βέβαια ή απόψεις. Μπορούμε να δούμε πώς θα πέλα. Δεν νομίζω να καταλήξουμε συμβαστική λύση. Είναι ακαθόδεστο το ζήτημα και στα πλαίσια του προπολογισμού. Ολόκληρο το άρθρο 55. Δεν με ε, λοιπόν που δεν έχουμε βρει ε, λύσει σε αυτό το πρόβλημα. Εξάλλου δεν μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Τροπολογία 12 για την άμεση στήριξη του προπολογισμού. Συζήτησα χτες ε, με τους προσώπους του ΕΛΚ, ε, διότι είχαν ανησυχίε για το άρθρο 3, για την εποπτεία, την παρακολούθηση μπορώ να την αντικαταστήσω με προφορική τροπολογία. Να διαγράψω το monitoring απλώς και να παραμείνει ε, έχει το κείμενο. Στην πρώτη τελευταία γραμμή διαγράφουμε το monitoring. Δεν πρόκειται για θεσμοθέτηση οποιοδήποτε πράγματος, απλώς διαγράφουμε το monitoring και το κείμενο παραμένει ακέραιο. Ελπίζω έτσι να λυθεί αυτό το ζήτημα της τροπολογίας 11. Κατά τα λοιπά θα συμπεριλάβω τα σχόλιά σας και έχω και μία πρόταση για την τροπολογία των φιλελεύθερων. Ένα λεπτάκι να την βρω. για τη διαφάνεια, όχι για τους δικαιούχους αυτούς, τους που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση, αλλά και τι την κάνουν τη χρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να δούμε. Ε, αυτά για τον προπολογισμό των εξωτερικών υποθέσεων στο τμήμα 4, έτσι, αλλά δεν θα υπάγεται στο τμήμα 4 αυτή η διάταξη. Είναι περίεργο τώρα να αναφερόμαστε λεπτομερώς σε αυτή τη χρηματοδότηση. Θα γίνει πιο γενικόλογη διατύπωση και ε, μήπως θα μπορούσατε να δεχτείτε την, ε, το να βγει αυτή η διάταξη από το τμήμα 4. Αν το δεχτείτε, μπορώ να ε, δεχτώ όλες τις υπόλοιπες ε, τροπολογίες. Οι σκιώδεις εισηγητές έχουν το λόγο τώρα, εάν το επιθυμούν. Κύριος Νεΐνσκι. Η κυρία Νέγινσκη, και συγγνώμη για την προφορά. Κυρίες αλλά και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το τόσο σημαντικό αυτό σχέδιο έκθεσης που νομίζω ότι θα μπορέσει να μας φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκαμψία στη διαχείριση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, προϋπολογισμού και φυσικά και καλύτερη λογοδοσία στα θέματα αυτά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε καταρχήν το θέμα της διαχείρισης των νεωστή ιδρυθέντων καταπιστευμάτων και επίσης τη διαχείριση του διοικητικού προϋπολογισμού των εξωτερικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπα και στην προηγούμενη συζήτηση, πιστεύω ότι τα καταπιστεύματα θα πρέπει να τυχάνουν διαχείριση μόνο από την Κομισιόν, επειδή είναι ένας νέος μηχανισμός, θα πρέπει να να την χάνουν ε, προσεκτικού ελέγχου από την Κομισιόν και να συμπεριλαμβάνονται στην απαλλαγή του προϋπολογισμού της Κομισιόν. Εμείς φυσικά ως Κοινοβούλιο δεν έχουμε τον ίδιο έλεγχο πάνω στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα ταμεία της. Εξάλλου θεωρώ απαράδεκτο ότι ο διοικητικός προϋπολογισμός των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης μπορεί να ξαναδοθεί στην Κομισιόν. Γιατί με τον τρόπο αυτό χάνουμε κάθε δυνατότητα ελέγχου και διαχείριση του προπολογισμού των αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούμε περισσότερο χάο από ό,τι ήδη υπάρχει. Ω Ευρωπαϊκή Ένωση εμεί δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια ισχυρή και στεναρή υπηρεσία εξωτερική δράση αν κάποιε από τι ευθύνε αυτή τη υπηρεσία θα τι επομιστούν άλλα θεσμικά όργανα. Αυτά λοιπόν τα θέματα που θέλουμε να υπογραμμίσουμε Αυτά εξ ονόματος του ΕΛΚ. Καλά λέει ο πρόεδρος. Άλλες ε, παρατηρήσεις. Εάν όχι, ευχαριστώ την κυρία Μπραντνερ και την κυρία Νέισκη και έχουμε κλείσει το σημείο αυτό. Ακολουθεί η έκθεση του κυρίου Σάριου Σπόλσκι, επικεφαλής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι εδώ ο κύριο Άιρου, ούτε ο κύριο Βόλτ και πρέπει να διακόψουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την κατανόησή σας. Δέκα λεπτά διακοπή. Ten minutes. <laughs> We have no chance anyway. Bene, il relatore è arrivato. Ξαναρχίζουμε. Όπως και κάθε χρόνο, από τις 27 έως το 30, έλαβε χώρα η Ανοιξιάτικη Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. 260 κοινοβουλευτικοί έλαβαν μέρος από τα διάφορα κοινοβούλια των χωρών του ΝΑΤΟ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπήθηκε από μια χωριστή αντιπροσωπεία και στη Βάρνα η αντιπροσωπεία μας απαρτιζόταν από πέντε μέλη, τον κύριο Σάιρους Φόλσκι, Πάσκου, Ριέρα Μαδουρέλ, Τάνοκ και Γιάτεν Μάκη. Και επειδή ήταν παρόν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Άμυνας και των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλγαρίας επίσης, και τα θέματα τα οποία ήταν τα κύρια ζητήματα που συζητήθηκαν στη Βάρνα ήταν η Αραβική Άνοιξη, τα θέματα του Αφγανιστάν, η νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ και η κυβερνο... Κυβε... κυβερνοάμυνα. Ο εισηγητής μας σας Βότσκι μπορεί να λάβει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δώσατε εσείς τα δεδομένα της κατάστασης, οπότε εγώ θα κάνω την αποτίμηση. Η αντιπροσωπεία μας προς την ε, ε, Επιτροπή Πολιτικής ε, Οικονομικών Επιστήμης και Τεχνολογίας. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ε, μας παρουσίασαν τις νέες στρατηγικές έννοιες, ε, κυρίως από βολγαρικής σκοπιάς, την άνοδο της Εκείνας, τις αραβικές επαναστάσεις, Λευκορωσία, και οι έσχατες στο Πακιστάν και οι επιπτώσεις που έχουν στην περιοχή του Αφγανιστάν. Στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας οι συζητήσεις στράφηκαν γύρω από την ομαδοποίηση και κατανομή των πόρων λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν ε, τα κράτη ε, Παρουσιάστηκε και μια ειδική έκθεση για τις σχέσεις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κυρία Μελίνε για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ βάσει της νέας στρατηγικής σύλληψης και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ιδιότητα του επιχειρησιακού εταίρου. Η υπέρβαση λοιπόν των φραγμών της συνεργασίας ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, αμοιβαία επωφελή συνεργασία των δύο. Η συγκήτρια αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες συνθήκης Λισαβόνα και τα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θέση εφαρμογή του πολιτικού οράματο. Επίση η συγγήτρια μίλησε για τι ε, ε, τρέχουσε στρατιωτικέ ελλείψει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, για την κρίση τώρα και τι επιπτώσει, καθώ και την ε, μικρότερη στήριξη τη κοινή γνώμης για τι ιδιωτικοποιήσει. Αναφέρθηκε η συγγήτρια στην Γάλλο-Βρετανική Συμφωνία του Νοεμβρίου για τη στρατιωτική στρατιωτική συνεργασία. Επίσης ήταν επικριτική σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. The plenary sitting uh, counted in Dalia, as you said, NATO Secretary General Στη Γενική Συνέλευση είχαμε και τον Γενικό Γραμματέα Ρασμούσεν, τον Υπουργό Αμήνη ε, της Βουλγαρίας ε, και τον Γενικό Διοικητή των Επιχειρήσεων ε, του ΝΑΤΟ στη Λιβύη. From the perspective of the previous... Ε, σε σχέση με τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές ε, συνελεύσεις κατά τη διάρκεια της, ε, αυτής της θητείας και συγκεκριμένα την τελευταία στη Βάρνα, σε σύγκριση με αυτές λοιπόν είμαι μάλλον απεσιόδοξος. Υπήρξε μια ολιγορία, μια έλλειψη ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια σανθήκαμε την Μάρλιν Ολμπράιτ και το επιτελείο της γενικότερα θα έλεγα ότι υπήρξε μία έλλειψη σεβασμού και ένα, μία διαφορία. Ε, εγκάρσια συζητήθηκαν σε όλες τις επιτροπές ε, τα ζητήματα. Επίσης μιλήσαμε για την ενιαία εντολή για την προστασία των, ε, στη Λιβύη Υπήρξαν κάποια ερωτηματικά για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, προστασία λοιπόν των πολιτών της Λιβύης, αλλαγή του καθεστώτος, χρονοδιάγραμμα για την λήξη των επιχειρήσεων, για την πυραυλική άμυνα, ε, μιλήσαμε για την πυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ και τη συνεργασία με τη Ρωσία. Αν η Τουρκία δεν θέλει να συμμετάσχει ε, στη δομή του συστήματος. Ε, η Βουλγαρία θα ε, υποδεχόταν ευχαρίστως στο δεύτερο ραντάρ Υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα, το σύστημα του ΝΑΤΟ και το σύστημα της Ρωσίας και θα μπορούσαν, είναι μια εναλλακτική λύση, να αναπτυχθούν εκ παραλλήλου αντί να έχουμε ένα ενίο σύστημα. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, πάντως αυτά ήταν τα βασικά συμπεράσματα για την πυραυλική ασπίδα, για το Αφγανιστάν. Στο ΝΑΤΟ έχουμε 132.000 στρατιώτες, ε, και μέχρι στιγμής 2.500 ε, νεκρούς με τον θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ε, ορισμένοι έκαναν έκκληση για την επιστροφή των στρατευμάτων και ακούστηκαν επικρίσεις για την αδιάκριτη θανάτωση αμάχων λόγω των επιθέσεων, κάποιων επιθέσεων του ΝΑΤΟ και υπήρξαν εκκλήσεις μέχρι το 2014 να έχουν αποσυρθεί όλα τα στρατεύματα για το Αφγανιστάν. Αυτά. Ε, ε, ε, για τη νέα στρατηγική έννοια μιλάμε για την συνολική ισορροπία της, του άρθρου 5 της συνθήκης της Ουάσιγκτον. Συζητήθηκε το θέμα της κυβερνοεγκληματικότητας, κυβερνοασφάλειας. Η Βουλγαρία κρίνει ότι θα πρέπει βάσει των εφεδρικών σχεδίων για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο για τις Βαλτικές χώρες να αναθεωρηθεί για την κυβερνοάμυνα τώρα είναι η υψηλή προτεραιότητα για τον ΝΑΤΟ ήδη από το 2007 ε, λόγω των κυβερνοεπιθέσεων ε, κατά της Εστονίας ε, υπάρχει το νέο ερευνητικό κέντρο στο Τάλιν και η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους συμμάχους αυτά είναι τα νέα στοιχεία αλλά υπολείπεται σοβαρή δουλειά, αλλά ε, χρειάζονται όμως ειδικέ προδιαγραφές. Οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν προτεραιότητα σε αυτήν την ε, σύνοδο. Ε, υπήρχε μια διάσπαρτη εντύπωση ότι στις επιχειρήσεις της Λιβύης φάνηκε αδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, και παρά τον ε, σεβασμό και τις καλές σχέσεις που συνήθως έχει το ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις διάφορες συναντήσεις ε, συναντήθηκα με τον Dr. Κάρλ Λάμπερς, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, ο οποίος μου είπε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Τον προσκάλεσα σε μια συνεδρίαση μετά το καλοκαίρι στις Βρυξέλλες. Έγινε δεκτή η πρόσκληση. Τώρα θα δούμε πώς ακριβώς θα το χειριστεί. Ε, στα πλαίσια της ενίσχυσης των σχέσεων ε, της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαμε ότι θα πρέπει να προβληθεί ο ρόλος του ΝΑΤΟ κυρίως στο Βουκουρέστι τον Οκτώβριο στην 57η Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, όπου ίσως προκύψουν και νέες προτάσεις. Grazie al Ευχαριστώ τον κύριο Σάριους Βόλσκι ο οποίος είναι ο εισηγητής. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να λάβει τον λόγο, ίσως. Ο κύριος Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Σάριους Βόλσκι, κάποιες ερωτήσεις για την τόσο ενδιαφέρουσα σας έκθεση. Συζητήθηκε το θέμα του Βερολίνου συν στην ε, Σύνοδο του ΝΑΤΟ δηλαδή ακριβώς το θέμα της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και η αντιμετώπιση του τουρκικού βέτο. Γιατί θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία στρατιωτικής και πολιτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ σε περιπτώσεις όπως το Αφγανιστάν. Γνωρίζουμε ότι το βέτο του, της Τουρκίας δημιουργεί προβλήματα για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Με ενδιέφερε να ξέρω αν υπήρξαν συζητήσεις για το θέμα αυτό για το να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το βέτο το οποίο δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης για το αντιπυραυλικό σύστημα το οποίο θέλει να εγκαταστήσει το οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ξέρουμε ότι η τσεχική δημοκρατία ε, βάσει, μέσω του Υπουργού Βόντρα δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για το σύστημα αυτό να εγκατασταθεί στο έδαφος της γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει επαρκής δέσμευσης από την πλευρά των Αμερικανών για το σύστημα αυτό στην Τσεχία. Θα ήθελα να ξέρω επίση αν υπήρξε κάποια συζήτηση για το θέμα αυτό. Και επίσης αν υπάρχει κάποια πρόταση να συμμετάσχει και η Ρωσία σε συζητήσεις της ε, ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να λάβουν μέρος σε μια κοινή συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ όλοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Τάνοκ. για τη κοινοβουλευτική συνάλευση του ΝΑΤΟ. Ε, κάτι θα πω. Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει ο κύριο Στάνοκ. Κάτι θα βρω να πω. Στη, αυτή που είναι στη Βάρνα, ήμουν εκεί ως ε, πρώτος αντιπρόεδρος στην αντιπροσωπεία αυτή. Ήταν ε, ενδιαφέρουσες μέρες. Φοβάμαι ότι εγώ δεν ήμουνα ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ε, ακόμα κάπως ε, αλαζονική αντιμετώπιση που είχαν εναντίον μας οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, ενώ εμείς συμμετέχουμε περισσότερο από αυτούς στις συζητήσεις και κάνουμε πιο πολλή δουλειά. Είμαστε πιο επιμελείς στην εργασία μας και συμμετέχουμε πλήρως στις συζητήσεις. παρόλα αυτά μας ανθυποβλέπουν οι εθνικοί κοινοβουλευτικοί. Ίσως είναι ένα πολιτιστικό χάσμα το οποίο κάποτε θα γεφυρωθεί Συζητήσαμε φυσικά για το Αφγανιστάν εν λεπτομερία, για τα δρόμενα στη Λιβύη, για τον κίνδυνο επικαλύψεων στον το, στο χώρο του κέρατος της Αφρικής, στην Σομαλία και άλλες περιοχές. Όλα αυτά τα διάφορα θέματα λοιπόν έτυχαν τη συζήτηση. Υπήρξε μια σύνοδος η οποία ήταν ειδικά αφιερωμένη στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, <clears throat> αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ρόλος του σε όλα αυτά. Από την άποψη αυτή ήταν μάλλον αξιοθρύνητη αυτή η συζήτηση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες, να πιέζουμε τους εθνικούς κοινοβουλευτικούς και να τονίσουμε ότι μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα και είμαστε εκεί για να παίξουμε μαζί τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν συζητήθηκαν τα βασικά προβλήματα στη Βάνα. Ίσως με την αφορμή αυτής της συζήτηση τώρα θα μπορούσαμε να το θέσουμε. Είναι το θέμα των προβλημάτων του ΝΑΤΟ. μια ολοένα αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα ευρωπαϊκά σκέλη σε εισαγωγικά του ΝΑΤΟ και της ΕΙΠΑ. Ο κύριος Γκέιτς έκανε πολύ σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τις ανεπάρκειες του ΝΑΤΟ Και από την άλλη έχουμε και την απογοήτευση των Ευρωπαίων εταίρων για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρήσει ένα κλίμα ειρήνευσης με τη Ρωσία, είπα. Έχουμε λοιπόν πλέον χρόνο για να συζητήσουμε τα κύρια προβλήματα και όχι για αυτά τα οποία συζητήθηκαν στη Δάνα. Λίζεκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή αν κατά τη διάρκεια της συνόδου στη Βάρνα συζητήθηκε το θέμα της γεωργίας από δύο πλευρές. Πρώτον, το θέμα της κατοχής κάποιων περιοχών της Γεωργίας από το Ρωσικό στρατό και δεύτερον, στο πλαίσιο των προθέσεων της Γεωργίας να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Δεύτερη ερώτηση. Έγινε κάποια συζήτηση για την ε, ε, στρατιωτικοποίηση, την τόσο επικίνδυνη στρατιωτικοποίηση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και τρίτον, θα ήθελα να πω πως αν ο πρόεδρος Λάμες ερχόταν στο Κοινοβούλιο, καλό θα ήταν να συναντηθεί και με τη δική μας την Επιτροπή. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Θέλει να προσθέσει κάτι ο εισηγητής. Thank you. But Ευχαριστώ. Να απαντήσω στον Μπροκ πρώτα, αν και είναι απασχολημένος με τη Φραγκίσκα. Ζηλεύεις, θα του λέει ο Μπροκ. Για το Βερολίνο Plus, Βερολίνο Συν, τίποτα καινούριο δεν ακούστηκε τώρα για την Τουρκία μέσω της πιθανής ικανοποίησης κάποιων ετοιμάτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξοπλισμών. Αυτά όλα βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η ίδια παρατήρηση την οποία είχα κάνει στα πλαίσια της πρώτης συνάντησης εδώ και λίγα χρόνια στο Εδιμβούργο εξακολουθεί να ισχύει. στην ουσία μας αντιμετωπίζουν όπως το κοινοβούλιο των κάποιων απόμακρων περιφερειακών περιοχών. Κάποιοι από εμά φυσικά προσπάθησαν να είναι υπερδραστήριοι, αλλά σε επίπεδο πρωτοκόλλου δεν μας έδωσαν καν το λόγο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με το Ράσμουσεν δεν μας έδωσαν ε, τον ε, λόγο. Το ίδιο επίσης έγινε και στη συζήτηση με το αρχηγείο του ΝΑΤΟ για τη Λιβύη, γιατί είχαν μια εντελώς διαφορετική λογική σε επίπεδο πρωτοκόλλου. Παρ' όλα αυτά ήμασταν υπερδραστήριοι όπως είπα. Και το πρόβλημα είναι ότι οι συνάδελφοι από τα εθνικά κοινοβούλια ζουν σε ένα διαφορετικό κόσμο. άλλοι ασχολούνται με το ΝΑΤΟ, άλλοι ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δύο αυτοί τομείς δεν εφάπτονται και υπάρχει πρόβλημα να μας καταλάβουν και οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εδώ επανέρχομαι στο σημαντικό ψήφισμα των Μπροκ, Γκουαλτιέρη και τα λοιπά για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο πώς θα μπορέσουν δηλαδή το επίπεδο το κοινοτικό και το εθνικό κοινοβουλευτικό να έρθει σε επικοινωνία. Η αδυναμία του κοινοβουλευτικού συστήματος είναι ότι σε επίπεδο επιρροής είμαστε διακοσμητικοί. Σε επίπεδο συζήτησης βέβαια είναι χρήσιμο γιατί δείχνει ότι ειδικευόμεθα σε θέματα ασφαλείας αλλά κυριαρχείται η συζήτηση από τις εθνικές απόψεις. Δεν υπάρχει επίπεδο επεξεργασίας θέσεων τοϊκό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε βέβαια. Με το ψήφισμα Γκουαλτιέρη Μπροκ και άλλων. Έχουμε λοιπόν την θρηνητική αυτή τη στιγμή πιθανότητα επικοινωνίας με τα κοινοβούλια τα εθνικά, σε επίπεδο πάντα κοινοβουλευτικό εννοώ, αλλά η διακοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και οι στρατιωτικοί, το προσωπικό κτλ. αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πιθανό συμπλήρωμα αυτού του οποίου κάνουν και σαν διαπραγματευτή με τον οποίο αξίζει να συζητήσουν. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα κενό ανάμεσα στις δύο οργανώσεις, την Ένωση και τον ΝΑΤΟ, και σε σχέση με αυτά που είπε ο Λαντσμπέργκης υπήρξαν ε, πράγματι ομιλίες που έδειχναν ότι πολλοί ζουν σε διαφορετικούς κόσμους. Δεν τέθηκε θέμα αμερικανικής εμπλοκής, του ποσοστού της αμερικανικής εμπλοκής και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να οικοδομήσουμε πράγματι ένα ευρωπαϊκό πυλώνα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ, που μπορεί να είναι η ίδια η ΚΕΠΑ, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε καθόλου μα καθόλου ικανοί να το κάνουμε. Σε επίπεδο αριθμών γνωρίζετε ότι εδώ και 20 χρόνια η ευρωπαϊκή συμμετοχή ήταν 50%, τώρα έχουμε φτάσει στο 25% σε επίπεδο δαπανών. Οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν λοιπόν τους Ευρωπαίους δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά μας αντιμετωπίζουν σαν παράσιτα. θεωρούν ότι τα ευρωπαϊκά κράτη δεν θέλουν να συμμετέχουν, δεν έχουν τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, δεν έχουν πυρομαχικά κτλ. Η κατάσταση λοιπόν είναι σοβαρή. Τα πλαίσια επικοινωνίας λοιπόν ελείπουν και αυτό φάνηκε και στις αδυναμίες οι οποίες ήρθαν στην επιφάνεια στα πλαίσια της λιβικής περίπτωσης και σε σχέση με τον προϋπολογισμό της επιχείρησης και όπως τα είπε άλλωστε ο Γκέιτς. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τα κοινοβούλια των κρατών μελών έτσι ώστε το θέμα του ΝΑΤΟ να τεθεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό και όχι εθνικό. Γιατί πάρα πολλές ομιλίες εκπροσώπων κρατών μελών στην ουσία δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να επαναλαμβάνουν ξεπερασμένα επιχειρήματα. Τώρα για τη Γεωργία. Η Γεωργία ουσιαστικά δεν ήταν στη μέρησια διάταξη σε καμία περίπτωση. Παρά την αντίδραση του Νατοϊκού Συμβουλίου τον προηγούμενο Αύγουστο μετά από την ε, εισβολή όταν είχαμε συνεδριάσει εκτάκτος υπήρχαν εν πάση περιπτώσει αντιδράσεις. Τώρα φαίνεται ότι όλοι έχουν δεχτεί το status quo και το θέμα δεν επηρεάζει τις σχέσεις με τη Ρωσία. Η Γεωργία λοιπόν είναι ένα μη θέμα ουσιαστικά. Κάποια σχόλια εκτός μικροφώνου. Η Γεωργία λοιπόν είναι ένα μη θέμα επαναλαμβάνω και το δικό μου προσωπικό μήνυμα και σε επίπεδο μιλιών και σε επίπεδο διαδρόμων είναι ότι η συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν ήταν αποτυχημένη. Θυμάστε τον Γερμανό στρατηγό που διαμαρτυρήθηκε, επέστρεψε διαμαρτυρώμενος λέγοντας ότι αυτά τα οποία συνεισφέρουμε είναι λίγα και δεν τα εκτιμά το ΝΑΤΟ. Η Λιβύη είναι η τελευταία ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε. Η κατάσταση όμως διαψεύδει αυτό το μήνυμα. Δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και πολλές φορές ακόμα και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας οι εκπρόσωποι της χώρας στα διαφορετικά φόρα ε, λειτουργούν με διαφορετική λογική και γλώσσα. Επανέρχομαι πάντα στην έκθεση Μπροκ Γκουαλτιέρη σχετικά με την διάσταση της ασφαλείας. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή λογική, μια κοινή πολιτική κατευθυντήρια για τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Μας έχουν ξεπεράσει τα πράγματα στα ε, οικονομικά, ξέρουμε περί του χρεοστασίου του ελληνικού, λέει ο κ. Σταουσβόλσκι. Μας έχουν ξεπεράσει τα πράγματα και εμείς οι Ευρωπαίοι που έχουμε 2 εκατομμύρια στρατιώτες τυπικά, θεωρητικά, δεν είμαστε σε θέση να, να προσφέρουμε 40.000 κόσμο όταν αυτό χρειαστεί. Και αυτή είναι η αλήθεια, η πικρή αλήθεια για την Ευρώπη. Και είναι κρίμα που ισχύουν αυτές οι καταστάσεις, αλλά δυστυχώς και το ΝΑΤΟ και οι αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναθεωρήσουν την διάσταση ασφαλείας και άμυνας σε επίπεδο ε, θα έλεγα τυπικό έχουμε την ΧΕΠΑ. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει. Έχουμε στρατιωτική συνεργασία η οποία είναι ανύπαρκτη πιστεύουμε. Έχουμε υποτίθεται αντιπροέδρους σε υψηλό επίπεδο για τα εξωτερικά θέματα που ίσως υπάρχει αλλά καθυστερεί. Αυτό το οποίο περιμένουν οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι ασφάλεια και αν αποκαλυφθεί ότι στην περίπτωση που δεν έχουμε την δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε περίπτωση κρίσης, όπως δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και στην κρίση του ευρώ βέβαια, τότε θα σημάνει το τέλος της προσπάθειας που κάνουμε. Ο συνάδελφος Τάνοκ. Κάτι ξέχασα. Υπήρξε κάτι το οποίο ήθελα να πω και τώρα που το ανέφεραν επανήλθε στο πνεύμα μου Συμφωνώ με τον Γιάσεκ ότι υπάρχουν πολλές φραστικές δηλώσεις ε, θετικές για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συμπληρωματικότητα προς τον ΝΑΤΟ, αλλά γενικά η αντίληψη είναι πάρα πολύ αρνητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και για την περίπτωση του Αφγανιστάν, οι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EUPOL ε, έτυχαν επιθέσεων από ένα εστονό εθνικό βουλευτή. Η Βρετανία όμως ήταν η πιο αρνητική για την παρουσία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώ ο κύριο Πάσκου δεν είναι παρόν σήμερα. Ο κύριο Πάσκου μα είπε και εγώ το ε, διαπίστωσα για το συγκεκριμένο αυτό βουλευτή επειδή γίνονται συνεδριάσει με επί επίπεδου πολιτικών οικογενειών υπήρξαν από τους σοσιαλιστές, εθνικού βουλευτέ, ε, έντονες επιθέσεις για τους ε, ευρωβουλευτές και το ρόλο τους από ένα ε, Βρετανό εργατικό, ένα εξέχοντα Βρετανό εργατικό που είναι κανονικά ένας ε, λογικός άνθρωπος Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμω επετέφθη περίπου ανετίως κατά των Ευρωβουλευτών για τα θέματα αυτά και τους υπερασπίστηκε πολύ καλά ο κ. Πάσκου. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη εχθρικότητα των εθνικών βουλευτών, δυστυχώ με επικεφαλή του ε, Βρετανούς για την ανάμειξή μα σε οποιαδήποτε τέτοια ε, λειτουργία των κοινοβουλευτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μας επαναφέρει αυτό στο θέμα της αντικατάστασης της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ που συζητάει αυτήν ο κύριος Μπρόκ και ο κύριος Νταφ. Και το ερώτημα είναι αν μπορούμε να βρούμε ένα νέο modus operandi και η πρότασή του ήταν όχι 6 μέλη αλλά 10% όλης της ε, συνέλευσης, δηλαδή 15 μέλη θα μπορούσαν να είναι ευρωβουλευτές και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε και ένα μεγαλύτερο ποσοστό αν έχουμε την κατάλληλη συμβαστική λύση, αλλά αυτό εξαρτάται και από τη θέση του Κοινοβουλίου μας και των εισηγητών. Χρειάζεται όμως να κλείσουμε αυτό το κενό και ώστε να επιτευχθεί αυτό θα εξακολουθούμε να είμαστε σε ένα διέξοδο, αλλά ο κ. Πάσκου με πολύ γενναίο τρόπο υπεστήριξε τους ευρωβουλευτέ στην ομάδα της Σοσιαλιστική εκεί. Κάποιο άλλο θα ήθελε το λόγο. Το επόμενο θέμα πρόταση ψηφίσματος για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία ανάμεσα στη CFC και στην CSTP. Στην τελευταία συνάντηση προετοιμάσαμε μία πρόταση ψηφίσματος η οποία κατά κάποιο τρόπο μας οδηγεί στο να συνεργαστούμε με τα κοινοβούλια των κρατών μελών στα πλαίσια της παρακολούθησης των μορφών συνεργασίας σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσουμε στον πρόεδρό μας μια ξεκάθαρη εντολή. Η συζήτηση για τη συνεργασία την διακοινοβουλευτική στον τομέα της EFCP είναι το πρωτόκολλο 1. Το άρθρο 10 του πρωτοκόλου αυτού προβλέπει στην ουσία την δυνατότητα οργάνωσης συναντήσεων με τους συναδέλφους από τα κοινοβούλια των κρατών μελών για να συζητήσουμε τα θέματα της CFSP e και της CSDP. E that of arguing that any form of interparliamentary cooperation, including in this area, Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 9 πάντα του πρωτοκόλου πρέπει να υπάρξει μια πρώτη συμφωνία από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον τομέα λοιπόν της ΚΕΠΑ και της ΕΠΑ μας δίδει η συνθήκη την δυνατότητα παρακολούθησης αυτών των πολιτικών. Η παρουσία μας σε κάθε διακοινοβουλευτικό φόρουμ που ασχολείται με τέτοια θέματα θα πρέπει να αναλογεί στον θεσμικό ρόλο τον οποίο έχουμε σαν κοινοβούλιο οι διαπραγματευτές μας, οι κύριοι Μπρόκ, Γκουαλτιέρη και Νταφ. Προετοίμασαν ένα κείμενο το οποίο μοιράστηκε ήδη χθε, αλλά είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα. Βασίζεται στα προηγούμενα έγγραφα, ιδιαίτερα την έκθεση Αλμπερτίνη και Γκουαλτιέρη την οποία μόλις ψηφίσαμε. Αν μπορούμε να ψηφίσουμε για τα κείμενα αυτά, τότε το απόγευμα ο Πρόεδρος κ. Σταλμπερτίνη θα το καταθέσει προς την Ολομέλεια και η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, θα αποφασίσει να το συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Θα δώσω τώρα το λόγο σε αυτούς οι οποίοι συνεισέφεραν στη διατύπωση αυτή. Καταρχάς θα ξεκινήσω με τον συνάδελφο Χέρμαλ Μπρόκ. Μόνο μια παρατήρηση ω προσθήκη έχω να κάνω σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν και δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που παρουσίασε ο εισηγητή. Θα πρέπει να δούμε ότι στο θέμα αυτό υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ εθνικών κοινοβουλευτικών και ευρωπαίων κοινοβουλευτικών, αλλά ακόμα και μέσα στα εθνικά κοινοβούλια υπάρχουν αντιπαραθέσεις με αυτούς που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα και αυτούς που ασχολούνται με την ευρωπαϊκή πολιτική. Η ΚΟΖΑΚ ίσω μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά, αλλά η ΚΟΖΑΚ εξακολουθεί να είναι χώρο συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων και είναι περιορισμένη συμμετοχή των Ευρωβουλευτών. Στην διακοινοβουλευτική αυτή συνέλευση υπάρχει το σημείο 9 και στην τέταρτη παύλα αναφέρει ότι ο στόχος της συνεργασίας αυτής μεταξύ εθνικών και ευρωπαίων βουλευτών είναι να υπάρξει μια κοινή διαμόρφωση θέσης. Αυτό σημαίνει και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην είμαστε επομένως μόνο η 28η αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Επομένως υπάρχει η ανάγκη να υπάρξει και συμμετοχή στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης και στην γραμματεία. Όλα αυτά απαιτούν και μια συμβολή της πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας έχει δώσει δικαιώματα να απαιτούμε τη λογοδοσία από την υψηλή εκπρόσωπο και επίσης και δικαιώματα στο επίπεδο του προϋπολογισμού και επίσης και μια δυνατότητα ελέγχου σε σχέση με την διαχείριση των κρίσεων από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, στα θέματα στρατιωτικών ενεργειών η χρηματοδότηση εξαρτάται αποκλειστικά από αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εδώ <clears throat> υπάρχουν ορισμένα εθνικά κοινοβούλια που ζηλοτύπωστοι θέλουν να διατηρήσουν τα προνόμια τους έναντι των εθνικών τους κυβερνήσεων και από την άλλη μεριά υπάρχει το θέμα της ε, συμβολής και της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύνολη διαδικασία. Όλοι οι βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια φαίνεται ότι έχουν μια λαθασμένη εντύπωση για αυτά τα οποία περιλαμβάνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό το είδαμε και στην συνάντηση με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης, με την Τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Προεδρίας. Είναι απαραίτητο επομένως να υπάρχει μια σαφέστερη εντολή για την αντιπροσωπείες μας σε σχέση με τις αποφάσεις που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία με τους εθνικούς κοινοβουλευτικούς στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μια σαφή θέση στην αντιπροσωπεία μας ώστε το επόμενο εξάμεινο να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα θέματα αυτά, εφόσον θα είναι και η Πολωνία η οποία θα έχει την, Πολωνία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους Πολωνούς φίλους μας τη ΕΜΤ να κατανοήσουν λίγο καλύτερα, ίσως ότι είναι απαραίτητο να συνεργαστούν μαζί μας για μια καλύτερη συμβαστική λύση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλευτικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για μένα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις οι οποίες θα δημιουργούνται και επομένως παρακαλώ όλους τους συναδέλφους στην Επιτροπή μας να ασκήσουν και αυτή την απαραίτητη επιρροή ώστε να γίνουν δεκτές οι θέσεις μας. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν και όλα τα θέματα τα λεπτομεριακά τα οποία έχει προβάλει το Κοινοβούλιο με στόχο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Ο κύριος Γκουαλτιέρη δεν είναι παρόν. Κύριε Ντόφ, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη της απόψεως των ε, τριών βουλευτών. Μια απόψη η οποία προσπαθεί να ανοιχνεύσει και να στηρίξει τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου και αυτό με τον πιο δυνατό συστηματικό θα έλεγα τρόπο. Η προηγούμενη συζήτηση που έγινε για το ΝΑΤΟ δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην ΚΟΣΑΚ αλλά είναι κάτι το οποίο καλύπτει περισσότερο χώρο. το σύνολο της πολιτικής δραστηριότητας των κρατών μελών, των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Εκτιμώ λοιπόν την εμπιστοσύνη σας είναι σαφές ότι θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου, όχι γιατί είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι σε σχέση με το κοινοβουλευτικό μας επίπεδο, αλλά γιατί έχουμε σαν στόχο να βελτιώσουμε την ποιότητα της ΚΕΠΑ. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έρθει να συνδράμει το Συμβούλιο και η λύση η οποία προτείνεται από την ΚΟΖΑΚ δεν θα λειτουργήσει καλά ούτε για την ΚΟΖΑΚ γιατί αποκλείει ουσιαστικά τους ειδικούς των, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας στα διάφορα κοινοβούλια. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λειτουργήσει. Και εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τους ομιλητές σε τέτοιου είδους συναντήσεις και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ΚΟΖΑΚ. να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Μπούζεκ θα εκτιμούσε μια ξεκάθαρη καθοδήγηση από πλευράς μας και αντίστοιχα και από την Ολομέλεια. Γιατί ο κύριος Μπούζεκ είναι αυτός ο οποίος εκφράζει την γραμμή μας και μάλιστα και με την επερχόμενη Πολωνική Προεδρία. Η διαπραγμάτευση γι' αυτό δεν θα είναι εύκολη. Ελπίζω λοιπόν η Επιτροπή σήμερα το απόγευμα να δεχτεί την πρόταση αυτή και η διάσκεψη των Προέδρων να συμφωνήσει και αυτή έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η σημαντική διαδικασία. So next speaker, Mr. Tanak, please. Κύριε Τάνοκ, ναι, ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ κάπως έκανα μια έμεση αναφορά στο θέμα αυτό προηγουμένως. <clears throat> Γνωρίζω ότι σε τελική ανάλυση για τα εθνικά κοινοβούλια, ιδίως για τους Βρετανούς και τους ε, Γάλλους, είναι ότι εμείς θα πρέπει να παίζουμε το ρόλο μιας ακόμα αντιπροσωπείας με το ίδιο μέγεθος έξι βουλευτές δηλαδή όπως και οποιαδήποτε εθνική αντιπροσωπεία. Εγώ το ανέφερα στον Βρετανό επικεφαλή τη επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι ένα λογικό άτομο και δεν είναι αντιτιθέμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά προφανώ θα πρέπει να αντανακλά τι απόψει τη Βουλή των Κοινοτήτων. Καλό άνθρωπο είναι παρόλα αυτά, μπορούμε να συνεργαστούμε και του είπα ότι έξι βουλευτέ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αρκούν για μα. <clears throat> και για το ποσοστό το οποίο αυτό θα μπορούσε να δεχτεί το 10% ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στέλνει 15 βουλευτές από 150. Εγώ θα έλεγα ότι η ομάδα μου θα μπορούσε να δεχτεί κάτι αυτού του επίπεδου. Με, του εξής ότι με έξι βουλευτές οι Βρετανοί οι ευρωβουλευτές δεν θα εκπροσωπούνται. Επομένως θα ήταν σαν να απαρνείται το ίδιο του το κόμμα. Επομένως ο Βρετανός αυτός ε, επικεφαλής αντιπροσωπείας είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις, μπορεί να αποδεχθεί αντιπροσωπείες. Εγώ έκανα μια διαφορετική πρόταση, αν τα 27 οι 27 βουλευτές είναι κάπου 7.300 και είμαστε εμείς 750. Όχι, είναι 7.700 οι εθνικοί βουλευτές και εμείς είμαστε 750 και βγαίνει αυτό 12% λέει ο κύριος Σταρό. Είναι περίπου 12% το ποσοστό των ε, η αναλογία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν έχουμε λοιπόν περίπου 20 βουλευτές με δυνατότητα ετήσιας αναθεώρησης, μπορούμε ίσως να βρούμε μια συμφωνία, γιατί δεν θέλω να καταλήξουμε σε ένα διέξοδο και επίσης να ζητήσουμε ένα μη, πραγμα... μη ρεαλιστικό αριθμό 30-40 όπως έλεγε ο κύριος Ντάφ, πούμε να είμαστε περίπου το 25% όλη τη συνέλευσης. Ο φόβος μου ο οποίος έχει επαληθευθεί από την, από την πείρα του παρελθόντος είναι ότι δεν θα έρχονται οι, εθνικοί, οι εθνικοί βουλευτές. Δεν θα έρχονται καταρχήν οι ευρωβουλευτές γιατί έχουμε μια εκατοντάδα εθνικών βουλευτών και είμαστε τρεις και ο κούκο εμείς και αυτό μα κάνει να γελιοποιούμεθα. Δεν μπορούμε λοιπόν να διεκδικούμε το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο της συνέλευσης όταν εμείς δεν θα μπορούμε να είμαστε παρόντες σε αυτές τις συνεδριάσεις. Αν κρατήσουμε ένα μικρότερο αριθμό και μπορούμε να τον ε, αναθεωρούμε σε τακτικά διαστήματα αυτό θα είναι καλύτερο. Και το άλλο, το οποίο ξέρω από τους ε, Βρετανούς, εθνικούς βουλευτές, λένε ότι δεν πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι αυτό που δίνει τη γραμματεία και να καθορίζει τον, τρόπο συνεδρία, τον συνεδρίας, γιατί αυτό είναι ευρωπαϊκοποίηση της συνέλευσης. Η δική ε, θέληση είναι να γίνονται αυτά στα εθνικά κοινοβούλια με εκπεριτροπής προεδρίες ή με κάποιες διαδικασίες ad hoc όποιο κοινοβούλιο έχει μια άδεια αίθουσα παραδείγματος χάρη να γίνεται εκεί πέρα συνεδρίαση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε και εκεί μια συμβαστική λύση. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεδριάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσω οι ευρωβουλευτέ να χαίρονται που πηγαίνουν και σε άλλα κοινοβούλια. Δεν ξέρω ποια είναι η απόψη του Άντριου και του Έλμαρ για του αριθμού γιατί αν επιμείνουμε πολύ για την αριθμητική μας παρουσία δεν θα πετύχουμε τίποτα. Σάριος Βόλσκι. Ευχαριστώ. Λόγω της ιδιαιτερότητας της ΚΕΠΑ και της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, γιατί γι' αυτό έχουμε δύο ακρονίμια, χρειαζόμαστε τα δύο κοινοβουλευτικά επίπεδα, όπως είπαμε σε προηγούμενες συζητήσεις. The main question is not how many. Το βασικό ζήτημα δεν είναι πόσοι θα μας προσωπήσουν, όπως λέει ο Τσάρλς, αλλά ποιοι. Ποια θα είναι η σύνθεση, ποιοι θα έρθουν από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από πού θα έρχονται. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω αυτά που ήδη έχω πει. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι στην ΚΕΠΑ. ΝΑΤΟ, και οι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβουλία των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και οι υπόλοιποι στο η ΚΟΣΑΚ δεν είναι το ιδανικό βήμα γιατί θεωρώ ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται καν τη φύση του προβλήματος. Γιατί όχι ΚΟΦΑΚ. Να σας θυμίζω και τι είναι ΚΟΦΑΚ. Ε, είναι η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, σε αυτή την συνεδρίαση ήμουν Γι' αυτή σας έλεγα προηγουμένως. Από την εμπειρία μου θα έλεγα ότι η ΚΟΦΕ που έχει μια ικανοποιητική εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων προσπαθεί να επανεφεύρει τον τροχό. Θυμάμαι ένα βουλευτή από τη Βουλγαρία, δεν ήταν υπουργό ε, άμυνα τη Βουλγαρία. Πώ τον λέγανε, Σάλμον Πάση άρχισαν να συζητούν καλή την πίστη, επανεφεύροντας το κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει. Όταν τους το είπαμε έμειναν άναυδοι. Ήθελα να κάνουν κοινέ αποστολέ, αποστολέ παρατήρησης, να πηγαίνουν πέρα, δόθε και να ε, επανειδρύσουν κάτι που ήδη υπάρχει. Δεν Είναι σημαντικό λοιπόν όχι μόνο ο αριθμός, αλλά και το ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα μας εκπροσωπούν. Δεν συμφωνώ με την, τον ενδιασμό του Τσάλς ε, Τάνοκ. Το σημαντικό είναι ποιοι θα έρθουν από τα διάφορα τμήματα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αν θέλουμε να έχουμε διπλή ιδιότητα, εντάξει, δηλαδή θα ασχολούμαστε με τι εξωτερικές υποθέσεις, με τι σχέσει ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να στείλουμε κάποιον από τη γραμματεία, ε, διότι οι άλλοι αγνοούν την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία όντως ε, και αυτό απορρέει από την δυσάρεστη κατάσταση. Ε, δηλαδή τα κοινοβούλια έχουν τα συντεχνιακά εγωιστικά ε, συμφέροντά τους τα οποία υπερασπίζονται και είναι κοντόφθαλμοι, δεν έχουν όραμα δεν καταλαβαίνουν πόσο κατεπήγον είναι το ζήτημα γιατί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ως προς τις επιχειρήσεις επιτόπου δεν θα καταφέρουμε τίποτα εάν δεν έχουμε μια συγχώνευση του ευρωπαϊκού και του εθνικού επίπεδου έχουν τις ευαισθησίες τους. Όλοι πρέπει να υπερβούμε τις ευαισθησίες μας. Perhaps because no name of... Κανείς δεν, είναι από... Κανείς δεν αναφέρεται μέσα στην έκθεση από την ΚΟΦΑΚ. υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων με του οποίους μπορείτε να συζητήσετε και να κάνετε από κοινού μια παιδαγωγική προσπάθεια είναι μάλλον οι άνθρωποι της ΚΟΦΑΚ. Αν ήταν εγώ να αποφασίσω για την ε, εκπροσώπηση, όποια και αν είναι η σύνθεση, είτε μιλάμε ε, για ε, εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να προέρχονται οι άνθρωποι από τι αντιπροσωπείε για τον ΝΑΤΟ, από τι Επιτροπέ Εξωτερικών Υποθέσεων κτλ. φυσικά δεν πρέπει να μπούμε στα δικά τους τα χωράφια, θα πρέπει να σεβαστούμε τις ευαισθησίες τους, αλλά Σίγουρα θα πρέπει να έρθουν κάποιοι από τι Επιτροπέ Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν πρόκειται μόνο για την εξωτερική πολιτική. Σίγουρα δεν είναι η Κόζακ το ιδανικό βήμα και σίγουρα δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι αυτοί που ειδικεύονται για τον ΝΑΤΟ αλλά δεν ξέρουν τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστροφο. Έτσι, αυτοί που γνωρίζουν τα περί Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούν ακόμη ότι υπάρχει και πάει επειδή διαβάζουν τις εφημερίδες αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται ουσιαστικά στον πραγματικό κόσμο. Ευχαριστώ συνάδελφε η κυρία Μπέντερ. E Πρώτα η σας ευχαριστώ. Θα ήθελα εν συντομία να πω ότι υποστηρίζουμε την προσέγγιση του κυρίου Μπροκ και του κυρίου Γκουαλτιέρη και φυσικά τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά με τους εθνικούς μας κοινοβουλευτικούς και παρακολουθούν το θέμα αυτό και συμφωνώ ιδιαίτερα με την παράγραφο 2. Και απλώς αυτό ήθελα να πω ότι είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζω απόλυτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αντικαθιστώ τη συνάδελφο την κυρία Λόσινγκ, η οποία δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα στη συνεδρίαση. Η δική, μου, μας παρατήρηση, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι μέσα από αυτή την διακοινοβουλευτική συνέλευση και γενικότερα από τη συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, αυτό που πρέπει να προσεχθεί και θα επιμείνουμε ακόμα περισσότερο είναι να διατηρηθεί για να μην πω να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τα ζητήματα όπως γνωρίζετε <clears throat> εξωτερικής πολιτικής και άμυνας είναι ακόμα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δυστυχώς δεν κατάλαβα ορισμένες έτσι τις εξέλαβα απαξιωτικές διαπιστώσεις σχετικά με το επίπεδο και την αντίληψη των εθνικών κοινοβουλίων Υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα, σας λέω, στα οικονομικά θέματα με το Ευρωπαϊκό Εξάμενο αφαιρείται ουσιαστικά και η δυνατότητα να χαράσουν οικονομική πολιτική τα εθνικά κοινοβούλια και στο επίπεδο που συζητάμε πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Με αυτή την έννοια λοιπόν ε, και σύμφωνα με το πρωτόκολλο το πρώτο της Λισαβόνας και τα άρθρα 9 και 10 εμείς πιστεύουμε πως ε, πρέπει να υπάρξει κοινοβουλευτικός έλεγχος της ΚΕΠΑ και της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και πρέπει να διανεργείται από τα Εθνικά Κοινοβούλια και βεβαίως και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τους εξής όρους, και αυτό θα ήθελα να τονίσω αγαπητοί συνάδελφοι κύριε Πρόεδρε, η διακοινοβουλευτική λοιπόν συνέλευση πρέπει να έχει κατά την άποψή μας το νομικό δικαίωμα να αρνείται ή να αποδέχεται την κάθε δράση της ΚΕΠΑ και όλων των πολιτικών και στρατιωτικών αποστολών. Δεύτερο, η διακοινοβουλευτική συνέλευση που προδευλέπει το άρθρο 10 επαναλαμβάνω του πρωτοκόλου και που περιλαμβάνεται και στο ψήφισμα, στο σχετικό ψήφισμα, στη σχετική πρόταση, πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητάει και να έχει πληροφόρηση, να στέλνει παρατηρητέ στι αποστολέ τη ΚΕΠΑ και τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Από αυτή την άποψη θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ότι χρειάζεται να υπάρξει διαδικασία πλήρους κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η οποία κατά την άποψή μας δυστυχώς έγινε εκτελεστικό όργανο της ΚΕΠΑ. Και τρίτο, να υπάρχει δυνατότητα τα κοινοβούλια να ζητούν γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις από την Υπηρεσία, ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Τέλος, κατά την άποψή μας, θα πρέπει η διακοινοβουλευτική συνέλευση να έχει το δικαίωμα να εγκρίνει δεσμευτικές γνώμες και ψηφίσματα, χωρίς όμως να περιορίζει τα εφιστάμενα δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων με οποιοδήποτε τρόπο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάμε με απαξιωτικό τρόπο σχετικά με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν έχω τάσεις περιχαράκωσης στο εθνικό, αλλά νομίζω ότι εκεί πρέπει να διατηρηθεί ο πραγματικός έλεγχος. Η συνεργασία μας δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των εθνικών κοινοβουλίων και βεβαίως ε, υπάρχει ένα ερώτημα από τη συζήτηση τι εννοούμε ποιος θα εκπροσωπεί τα εθνικά κοινοβούλια. Και το λέω αυτό επειδή η εκπροσώπηση των εθνικών κοινοβουλίων στη κοινοβουλευτική συνέλευση πρέπει να είναι αυθεντική. Αυτό σημαίνει ή δυνατόν εκπρόσωποι όλων των πολιτικών ομάδων, διότι συνήθως τέτοιες εκπροσωπήσεις είναι από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα τις δύο μεγαλύτερες κομματικές οικογένειες, με συνέπεια η εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων να μην είναι αντιπροσωπευτική όλων των απόψεων που υπάρχουν σχετικά με αυτά τα ζητήματα και, τα οποία, και οι οποίες απόψεις είναι απαραίτητες προκειμένου να υπάρχει η πραγματική αντίληψη και ουσιαστικός ρόλος ερετών οργάνων όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Α, ο Σάιλ Βόλσκι ξανά και μετά ξανά ο Νταφ. Πρώτος ο Σάιλ Βόλσκι, μετά ο Νταφ και μετά ο Μπροκ. Όπως σας είπα, λέει ο κύριος Σάιλ Βόλσκι, το επίπεδο των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων και το επίπεδο της ΚΟΖΑΚ δεν είναι το καλύτερο για να γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αντιπροσωπευτικό σώμα το οποίο να ψηφίζει και να λαμβάνει αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε τρεις Μαλτέζους θα έχουμε 30 Γερμανούς. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και προσπαθώ να πείσω και το ΣΕΙΜ, την Πολωνική Βουλή, στρέφομαι προς τον Κονζάτο εδώ, το οποίο δεν θα λέγεται διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών των Κοινοβουλίων Κρατών Μελών, αλλά των Προέδρων της των Επιτροπών Εξωτερικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκής Πολιτικής και θεμάτων του ΝΑΤΟ και Άμυνας. Δηλαδή εμείς θέλουμε ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτού του οργάνου μπορούμε ας πούμε να, να καλούμε δύο προέδρους, δύο αντιπροέδρους, τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας με τη συνέλευση του ΝΑΤΟ. Μπορούμε το φορμά να το φτιάξουμε. Δεν θέλουμε εμείς να φτιάξουμε ένα πλήρως αντιπροσωπευτικό σώμα το οποίο να βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο εμείς λειτουργούμε ή ε, πώς ε, ε, κάποτε είχε δημιουργηθεί και συνίστατο η ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή της, της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Ίσως σαν Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συγκαλέσουμε μια τέτοια συνάντηση χωρίς κανένα πρωτόκολλο, χωρίς κανένα τυπικό, απλά για να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τη συζήτηση αυτή στους προέδρους των κοινοβουλίων ή ε, στα χέρια της ΚΟΖΑΚ που δεν θα μας οδηγήσει το ταχύτερο δυνατόν σε αποτελέσματα. Οι ανησυχίες των Προέδρων όμως των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι κατανοούν την ανάγκη που υπάρχει και κατανοούν το κατεπήγον της ανάγκης αυτής. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε και να φανούμε δημιουργικοί και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με όσους μπορούν πράγματι να συνεργαστούν μαζί μας που μπορεί να μην εργάζονται στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς αλλά έχουν κοινέ ανησυχίες και αντιλήψεις για την κοινή εξωτερική πολιτική άμυνας και τα θέματα του ΝΑΤΟ. Αντίθετα από τη Φρανσίσκα η οποία δεν είναι εδώ τώρα πια, είπε ότι της αρέσει το σημείο 2. Για μένα δεν είναι λάθος, αλλά είναι κάτι το περιττό. Α, λέει χρειαζόμαστε διακοινοβουλευτική συνέλευση. Το σημαντικό είναι τρία. Λυπούμεθα για την έλλειψη συμφωνίας από την διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών. Αυτό μας έχει οδηγήσει σε ένα αδιόξελο. Για να φύγουμε από το αδιέξοδο θα πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαβούλευση. Εγώ θα πείσω την Προεδρία του Πολωνικού Κοινοβουλίου να υποστηρίξει και να προτείνει αυτή τη συνάντηση για να βγούμε από το αδιέξοδο. Για να μην συνεχιστεί αυτό το αδιέξοδο γιατί φοβάμαι ότι είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια αυτές τις δύσκολες εποχές. Ο κύριος Ντάφ έχει το λόγο. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που ελέγχθηκαν και ο Γιάσεκ έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι μια κομβική παράγραφος, η παράγραφος παριθμών 3, εκεί που έχουμε θεσπίσει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μετά από την ε, συνεδρία της Κόζακ στη Βουδαπέστη, οι περισσότεροι εθνικοί κοινοβουλευτικοί ήταν εκεί και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε υπάρξει συμφωνία και μπορούσε να υπάρχει μια ειδικευμένη εκδοχή της ΚΟΖΑΚ για τα θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής που θα το δεχόταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω πρέπει να το κάνουμε απόλυτα σαφές ότι δεν δεχόμαστε τέτοια αντιμετώπιση. Νομίζω ότι χρειάζεται χρόνος για να διαλύσουμε τις λανθασμένες εντυπώσεις και την άγνοια η οποία πλανάται πάνω από τα Εθνικά Κοινοβούλια σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε σχέση με την φύση της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Χρειαζόμαστε λοιπόν χρόνο για να ξανατοποθετήσουμε σωστά στο πλαίσιο αυτό το ΝΑΤΟ, να δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση και για να μπορέσει η κυρία Άστον και ο κύριος Φαν να καταγάγουν κάποιες επιτυχίες που δείχνουν ότι η ΚΕΠΑ πράγματι είναι λειτουργική και μπορεί να δώσει αποτελέσματα και μπορεί να προωθήσει και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον τομέα της άμυνας και των εξωτερικών θέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε επιτύχει ακόμα για να μπορέσουμε να δείξουμε σε όλους ότι λειτουργεί αυτή η πολιτική. Πιστεύω επομένω ότι οποιαδήποτε νέα μορφή διακοινοβουλευτικής συνεργασίας σε σχέση με τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να έχει και αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της γεωγραφικής και πολιτικής πολυμορφίας της Ευρώπης. Αλλά έχει δίκιο ο Γιάσετ ότι θα πρέπει να δώσουμε και τη δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό να εκφραστούν καλύτερα και να υπάρχει και ευρύτερη εμπειρογνωμοσύνη για τα θέματα αυτά, τα εξωτερικά και άμυνες, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Η Κοζάκ όμω από τη δική της πλευρά αποφάσισε να βάλει στο περιθώριο την Κόφακ ή Κόφαντ όπως λέγεται. του επικεφαλίζει των Επιτροπών Άμυνα. και θεωρεί ότι μπορεί να παίρνει αποφάσεις μόνη της χωρίς και μία διαβούλευση με τα ίδια τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα για την Πολωνική Βουλή να μπορέσει να ξαναδημιουργήσει ένα επικοδομητικό πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τα θέματα αυτά. Πρέπει παρόλα αυτά να προσπαθήσουμε να τους ενθαρρύνουμε, τους Πολωνούς να το κάνουν αυτό. Και πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό επιτυγχάνει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Για τον ε, Charles Στάνοκ θα ήθελα να του πω ότι η Βρετανική επιμονή να μην συνεδριάζουν μέσα στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα παράλογη και πεδαριώδης. Και φυσικά είναι και πολύ Γιατί το κόστος του να βρούμε τον κατάλληλο χώρο ο οποίος μπορεί να υποδεχθεί τον μεγάλο αριθμό των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης που είναι μια πολυμελής αλλά και πολύγλωση συνδιάσκεψη, το κόστος αυτό είναι πολύ μεγάλο πολλά εθνικά κοινοβούλια δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν, να βρουν τα λεφτά για να καλύψουν το κόστος αυτό. Οι Βρετανοί θεωρούν ότι οποιαδήποτε τέτοια νέα δομή θα πρέπει να συνεδριάζει στον γιους τους λήψιους, στο κτίριο του Συμβουλίου. Μα και αυτό είναι παραλογότερον του παραλόγου, γιατί ακόμα και εκεί δεν υπάρχει μια αίθουσα του μεγέθους που χρειαζόμαστε. Είναι λοιπόν πραγματικά λυπηρή η στάση των Βρετανών και η οποία καταρχήν απλώς καταδεικνύει την περιφρόνηση με την οποία ε, αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως αυτό δεν πρέπει να το πω ανοιχτά. Τώρα για το μέγεθος της αντιπροσωπείας μας δεν πρέπει να μας γίνει μονομανία ο αριθμός αυτός. Αλλά σίγουρα 6 είναι ένας γελίος αριθμός, ένας γελία χαμηλός αριθμός. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια εκπροσώπηση μονάχα. Το 20% του συνολικού αριθμού μελών που θα είναι 162 είναι 32, τέσσερις βουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμένα μου φαίνεται ότι αυτό είναι πολύ πρόσφορο, ιδίως όταν μπορούμε να έχουμε και 0,4 βουλευτού, ένα λίγο λιγότερο από το μισό ενός βουλευτού να συμμετέχει και σίγουρα αυτό ο αριθμό θα επιτρέπει να εκπροσωπείται και ένας Βρετανός συντηρητικός και ένα μέλος της ΓΚΟΕ. Ultimo Σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για αυτή την θέση. Αλλά πρέπει να γίνει σαφές ότι σε τελική ανάλυση θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ποσοστό 30 τα 100 Αν όμως ε, επιμείνουν τα εθνικά κοινοβούλια να είναι τέσσερις βουλευτές για κάθε ε, κράτος που συμμετέχει, θα πρέπει εμείς να επιμείνουμε να έχουμε 27 βουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο διαδικαστικό. Και επίσης εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει η Προεδρία να αποφασίζει που γίνεται που γίνονται συνεδριάσει. Σε πολλέ περιπτώσει οι αποφάσει αυτέ δεν λαμβάνονται στα Εθνικά Κοινοβούλια από τον πρόεδρο τη Βουλή, αλλά από του προέδρου των ε, πολιτικών ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι μια αντιπολίτευση δεν έχει πάντα τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μια, μια συνεδρίαση. Μόνο λοιπόν αν λάβουμε υπόψη την πολυμορφία των Εθνικών Κοινοβουλίων θα κατανοήσουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερα νόημα αυτό και θα πρέπει να αποφασίσουμε να αφήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια να μας πούν αυτοί ποιον θέλουν να στέλνουν στην ε, κοινοβουλευτική συνέλευση. Και έχω ακόμα δύο παρατηρήσεις να σας προσθέσω. Και το ένα που μου έχει υποδείξει ο κύριος Σάριος Βόλσκι είναι ότι δεν είναι σωστό να αφήσουμε τα θέματα αυτά στην ΚΟΖΑΚ. Και πρέπει τελευταία φράση στο σημείο 3 για αυτό το λόγο να, να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ΚΟΖΑΚ έχει το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις εξ ονόματος όλων. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Σάριους ότι δεν είναι ο κατάλληλο χώρο για τη λήψη αποφάσεων αυτό η Κόζακ. Αυτό είναι λοιπόν να διαγραφεί το τέλο τη παραγράφου 3. Και επίση πάλι στο σημείο 3 αναφέρεται στην Πολωνική Προεδρία κ. Μπροκ. Μία συμφωνία με τα Εθνικά Κοινοβούλια αυτό θα έπρεπε να διατυπωθεί λέγοντας μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε μπορούμε να τους επιβάλλουμε να καταλήξουν σε μια συμφωνία για μας. Πρέπει να πούμε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Uh, Μάλιστα, σίγουρα συμφωνώ με τον Έλμαρ για τη δεύτερη παρατήρηση που έκανε, διότι απηχεί αυτό που επιδιώκουμε αυτή η διατύπωση προτείνει. Για την επιτύξη συμφωνίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια για την πρώτη του πρόταση αυτή η ευγενής αναφορά στην ΚΟΖΑΚ ε, που πρότεινε, δεν νομίζω ότι θα χαρεί η ΚΟΖΑΚ. Στο τέλος της συνεδρίασης δε, είπαν ότι θα εξετάσουν περαιτέρω αυτές τις προτάσεις και θα ήταν πιο διπλωματικό από πλευράς μας ε, να ε, το αναγνωρίσουμε αυτό. Ευχαριστούμε και ο κύριος Μπρόκ για να κλείσει η συζήτηση. Συμφωνώ μαζί σας και οι δύο κατά κάποιο τρόπο δεν περάσαμε πολύ καλά στη συνάντηση του Βουδαπέστης. Νομίζω ότι το ευγενέστερο που μπορούμε να πούμε σε σχέση με την Κοζάκ είναι το να μην πούμε τίποτα. Σχετικά με τη Βρετανική αντιπροσωπεία και τη Γερμανική αντιπροσωπεία. καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Κοζάκη είναι αυτή η οποία θα πρέπει να αποφασίσει. Αλλά εμείς θα πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό δεν έχει σχέση με την Κοζάκ. Το ιδανικό ε, είναι να μην σχολιάσουμε την Κοζάκ και να μην πούμε τίποτα για αυτήν έτσι κι αλλιώς. Ο Έλμαρ Μπρόκ έχει πολύ περισσότερη εμπειρία με μένα. Είναι πιο όριμος από μένα θα συμφωνήσω μαζί του και θα μπορούμε νομίζω να διαγράψουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι της φράσης που αναφέρεται στην Κοζάκ. Κοιτάξτε, εννοεί ότι είμαι ανώτερος αλλά όχι γυρεότερος ελπίζω ο κύριος Νταφ. Λοιπόν σας ευχαριστώ λέει ο κύριος Πρόεδρος, διακόπτουμε μέχρι τις 11. Οπότε θα ξεκινήσει το Προεδρείο, το οποίο θα κρατήσει μισή ώρα μέχρι τις 11.30. Σας θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα το κείμενο αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία και μιας και δεν υπάρχει χρόνος για κατάθεση τροπολογιών, μπορούμε να ψηφίσουμε τροπολογίες παρά μόνο όμως προφορικές.